Please Καθίστε παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν, να καλωσορίσουμε σε αυτή την ε, έκτακτη κοινή συνεδρίαση τριών επιτροπών. Έχουμε εδώ την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. ΛΥΜΠΕ και Ντέβε. Είναι εδώ και ο κύριο Ντέβιντ Μακάλιστερ, πρόεδρο τη Επιτροπή ΑφΕΤΕ και ο κύριο Τεμπία Στόμπε, πρόεδρο τη Επιτροπή Ντέβε και εγώ. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και ας περάσουμε στις συνήθειες ανακοινώσεις για την έγκριση τη ημερησία διάταξη. Τώρα έχουμε κάποιε αλλαγέ στο σχέδιο ημερησία διάταξη. στο σημείο 4, σε σχέση με τι παρουσιάσει τη υπηρεσία εξωτερική δράση ε, και τη ΥΠΑ τη αρμοστία του ΙΕ για του πρόσφυγε. Ε, έχουν αντικατασταθεί από μια παρουσίαση του Μάικλ Κέλλερ, ο οποίο είναι αναπληρωτή Γενικό διευθυντή τη ΓΑΜΑ ΕΚΟ. Και τα σημεία 10 και 11 η σύναψη πρωτοκόλλου με την Ελβετία και το Λιχτενστάιν και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και της Νορβηγίας σε σχέση με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για ε, τη θέσπιση του κατάλληλου κράτους, του αρμόδιου κράτους για να εξετάσει το αίτημα ε, ασύλου που κατατίθεται σε κράτος μέλος στην Ελβετία σε σχέση με την πρόσφυση της Eurodac ε, για λόγους επιβολής του νόμου έχουν ανασταλεί, αναβάλλονται. Τώρα, σε σχέση με το γλωσσικό καθεστώς, έχετε όλες τις γλώσσες διαθέσιμες στη Δερμηνία, εκτός από κροατικά και ελλανδικά. Και περνάμε στην έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Ο Τόμα Ζεντόφσκι έχει διοριστεί εισηγητή για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία και ο Άντωνι Χουκ έχει διοριστεί εισηγητή για την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύνευση συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λευκορωσία για την έκδοση θεωρήσεων. Επίσης, έχουν διοριστεί εισηγητέ για τις γνωμοδοτήσει. Η κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα, γνωμοδότηση για την απαλλαγή. Γνωμοδοτήσει για την απαλλαγή, Αρκετέ. σε σχέση με όλου του οργανισμού. Αν συμφωνείτε, θεωρούμε ότι εγκρίνονται οι συστάσει αυτές από την Επιτροπή μας. Έχουμε για κάποια σημεία σε σχέση με την ε, κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικέ πράξεις. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον Πρόεδρο. Έχουμε μια κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και με την Επιτροπή Ανάπτυξης θα συζητήσουμε το θέμα του μηχανισμού της Τουρκίας ε, και την κατάσταση των προσφύγων από τη Συρία που βρίσκονται στη Τουρκία. Έχουμε παρουσίαση από τον κύριο Μασεποπόσκι, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΝΙΑΡ και παρουσίαση του κυρίου Μάικλ Κέλλερ, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ανθρωπιστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την ανταλλαγή απόψεων και στη συνέχεια στις 10 το πρωί θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Έλληνα Υπουργό που θα μας παρουσιάσει την κατάσταση του μεταναστευτικού ζητήματος στα ελληνικά νησιά. Κάτι πολύ ενισχυτικό. Ο κύριος Χρυσοχοίδης θα παρευρεθεί εδώ στις 10 για να συζητήσουμε το θέμα της κοινή ε, δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Αλλά πριν να ξεκινήσουμε, θα πρότεινα στους δύο συμπροέδρους, τον κύριο Μακάλιστερ, πρόεδρο της ΑΦΕΤ και τον κύριο Τόμπε, πρόεδρο της ΔΕΒΕ, αν θέλουν να μας πούν δύο πριν να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερικής διάταξης. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, Χουαν Φερνάντο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί έχουμε καθυστερήσει. Θέλω να πω ότι χαίρομαι που βλέπω ότι η πρακτική να έχουμε συναντήσεις για τις εξωτερικές πτυχές μετανάστευσης σε αυτό το κοινό φορμάτι συνεχίζεται. Όπως αναφέρεται, είναι σημαντικό να μην δουλεύουμε ο καθένα μεμονωμένα, αλλά να ενώνουμε τι δυνάμει μα στο Κοινοβούλιο όταν πρόκειται για τέτοια οριζόντια ζητήματα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν σήμερα το πρωί να ακούσουμε πώ έχει η κατάσταση, αλλά και το σχεδιασμό για το μέλλον δεδομένων ε, των. Την, ε, ε, ότι θα λήξει η δεύτερη δημοσιονομική περίοδος για το μηχανισμό για τους πρόσφυγες στα τέλη αυτού του έτους. Ο κύριος Στόμπε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πραγματικά θετικό ότι έχουμε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε. Έτσι λοιπόν, ε, αντί να κάνω κάποιες παρατηρήσεις τώρα, θα τα πω στο τέλος. Ωραία, ας περάσουμε με τις παρουσιάσεις. Καταρχήν το λόγο έχει ο κύριος Ποπόφσκι για 10 λεπτά. Κατόπιν θα μιλήσει ο κύριος Κέλλερ και κατόπιν θα ακούσουμε τους συντονιστέ δύο λεπτά τον καθένα και το πολύ για ένα λεπτό παρακαλώ να το θυμάστε. Για ένα λεπτό θα μπορείτε να πάρετε το λόγο. Γιατί στις 10 θα έρθει ο Έλληνας υπουργό, επομένως δεν ε, θα χρονοτριβήσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Οι σχέσεις ε, με την Τουρκία παραμένουν δύσκολες όπως γνωρίζουμε και συνεχίζει, υπάρχει συνεχής επιδείνωση της δημοκρατίας και του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και εξακολουθούν να υπάρχουν τεταμένες σχέσεις με κάποια κράτη-μέλη που μας ε, οδήγησε σε ένα de facto πάγωμα των διαπραγματεύσεων ε, για την προσχώρηση και για τον εξυγχρονισμό του Τελωνιακού Κώδικα. Είναι λοιπόν σε μια δύσκολη συγκυρία η σχέση μας ε, και λόγω της δράσης Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και πρόσφατα τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βόρεια Σύρια που έχει καταδικάσει δημοσίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επανέλθω σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ε, που είναι το πλαίσιο μέσο στο οποίο λειτουργήσαμε το 2016, Είχαμε πολύ αρνητική ρητορική από τον πρόεδρο της Τουρκίας ε, και την κυβέρνηση. Συνεχίζουμε όμως να σημειώνουμε καλή πρόοδο με την υποστήριξη των σύρων προσφύγων στην Τουρκία έχουμε ολοκληρώσει τον προγραμματισμό του πλήρους κονδυλίου των 6 ε, δισεκατομμυρίων. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τη διερμηνία, κάτι δεν δουλεύει. Σε ποια γλώσσα δεν ακούτε, γαλλικά. Τώρα ακούτε. Μάλιστα. Συνεχίστε παρακαλώ. Λοιπόν, ο προγραμματισμό του μηχανισμού για του προσφύγε στην Τουρκία, το εργαλείο των 6 ε, εκατομμυρίων που έχουμε, έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό σημαίνει ότι τώρα υλοποιούμε τις ε, δεσμεύσεις μας ε, σε σχέση με την δήλωση. Θα αναφέρω λεπτομέρειες σε λίγο. Έτσι λοιπόν παραμένουμε εκεί για να βοηθήσουμε τους Σύρους και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία και εργαζόμαστε για την ε, ασφαλή επανακατάσταση των προσφύγων προς την Ευρώπη. Τις τελευταίους δύο μήνες βέβαια είδαμε σημαντική αύξηση παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία. Αυτή τη φορά κυρίως ε, από το Ιράν, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και ζητήσαμε από τις ε, τουρκικές αρχές να μας υποστηρίξουν να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα στην Τουρκία για να εφαρμοστεί η δήλωση. Αυτό συζητήθηκε από τον Επίτροπο Αβραμόπουλο όταν ε, μετέβη στην Άγκυρα στις αρχές Οκτωβρίου. Ε, η Κομισιόν έχει προετοιμάσει μια σειρά μέτρων περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να δοθούν ως χρηματοδότηση μέσω της προταξιακής βοήθειας και του μέσου που συνεισφέρει στη σταθερότητα και την ειρήνη. Και έχουμε θέσει στόχο να βελτιώσουμε την ικανότητα της ακτοφυλακής Τουρκίας για να προβαίνει σε έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. Επίσης, συνεχίσουμε τη στήριξή μας ε, στην ε, Γενική ε, Κυβέρνηση για να έχουμε βελτίωση των υλικών επιδοχής και να βελτιωθεί η κατάσταση στα κέντρα κράτησης και Θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των μεταναστών και προσφύγων στην Τουρκία. Φυσικά, η στρατιωτική παρέμβαση, η στρατιωτική επέμβαση στη Βόρεια Συρία έχει περιπλέξει τα πράγματα. Ο πρόεδρος Γιούνκερ κατέστησε σαφέ ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, στην υποδομή για, την, ε, ε, για τον επαναπατρισμό των Σύρων στη βορειοανατολική Συρία δεν συζητείται καν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, δεν είναι βοήθεια σε περιοχές όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών. Ε, ε, νομίζω όμως ότι ο ε, Μίκαλ θα μιλήσει για τα θέματα αυτά, έτσι λοιπόν δεν θα με κρηγορήσω εγώ. Και σημειώνουμε φυσικά την πρόσφατη, το πρόσφατο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που καταδικάζει την επιχείρηση της Τουρκίας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για να χρησιμοποιηθεί, ε, δεν θα χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση. Ε, η Τουρκία αναφέρεται σε ασφαλή ζώνη, αλλά εμεί δεν χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο. Δεν πρόκειται για ασφαλή ζώνη. Πού βρισκόμαστε με την εφαρμογή για το μηχανισμό των προσφύγων στην Τουρκία. Πραγματικά ε, είμαστε ε, όπως το 90% του κονδυλίου των 6 εκατομμυρίων έχει προγραμματιστεί. Η δεύτερη δόση, επίσης σε ε, αυτό το χρόνο, έχουμε δώσει ε, από τα 3 τα 2,4 δις και Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι συμβάσεις ε, θα υπογραφούν μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. Θέλουμε να διατηρήσουμε τους ίδιους ε, τρόπους για την εφαρμογή, όπως και στο πρώτο στάδιο, δηλαδή εργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς, ε, τράπεζες, τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, της ΜΚΟ και δίνουμε κάποια άμεσες επιδοτήσεις στο Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, και κοινωνικών υποθέσεων στα Υπουργεία αυτά της Τουρκίας, όμως δεν είναι η δημοσιονομική υποστήριξη όπως τη γνωρίζουμε απλώς. Ε, καλύπτουμε το κόστος της τουρκικής διοίκησης ε, τις δαπάνες που έχουν προκύψει όταν χρηματοδοτούν προγράμματα για τους σύρους. Δηλαδή, ε, ουσιαστικά μιλάμε για το κόστος λειτουργίας κλινικών και σχολείων. Τα αποτελέσματα, κατά την άποψή μας, είναι ενθαρρυντικά είναι κάτι εφικτό, είναι κάτι απτό. Ξέρω ότι πολλοί από εσά στην προηγούμενη θητεία ταξίδεψαν στην Τουρκία. Έχουμε 90 προγράμματα που τρέχουν και θα φτάσουμε τα 120 μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους. 1,7 εκατομμυρία πρόσφυγες ε, λαμβάνουν στήριξη διαβίωσης. Έχουμε φτάσει σε έναν ε, καλό ε, αριθμό εγγραφή των παιδιών στο σχολείο. Πάνω από 500.000 ε, παιδιά πάνε στο σχολείο και Επίσης, ε, χρηματοδοτούμε την κατάρτιση και την εργασία των δασκάλων στο σχολείο για τα παιδιά των σύρων. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της υγείας. Έχουμε βοηθήσει να κατασκευαστούν 180 κέντρα για τους μετανάστες ε, και έχουμε εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό ιατρικού προσωπικού και υπάρχουν και δράσεις ε, που αφορούν την προστασία των ευπαθών ομάδων. Και τώρα δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική και οικονομική υποστήριξη, δηλαδή δημιουργία θέσεων εργασία για τι ε, οικογένειε των Σύρων, όπου και αν ζουν, δηλαδή ένταξη στην αγορά εργασία, επαγγελματική κατάρταση και απόκτηση προσόντων και η δεύτερη, ο δεύτερο νέο τομή προτεραιοτήτων και σίγουρα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε το θέμα τη παιδεία και τη υγεία. Το δεύτερο ε, τομέα προτεραιοτήτων λοιπόν είναι ε, η δομή των Δήμων. Έχουμε ήδη δώσει 380 ε, εκατομμύρια ευρώ για το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων και ύδατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τα μέσα του 2021 το αργότερο θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα προγράμματα και τα περισσότερα από τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν ε, ολοκληρωθεί. 2022 και 2023. Ε, παραμένει δύσκολη όμως η κατάσταση. Ο ρυθμός των ε, μεταναστών αυξάνεται στην Τουρκία. Υπάρχουν νέες αφήξεις και οι επιστροφές δεν είναι κάτι εγγυημένο. Έχουμε σαφή θέση για τις επιστροφές που σας ανέφερα πριν μας ε, προσέγγισε η τουρκική κυβέρνηση και ήθελε να μιλήσουν για το μέλλον και είπαμε ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε μια συζήτηση που να έχει νόημα, αλλά αυτό ήταν πριν να ξεκινήσει η στρατιωτική επέμβαση. Και είναι δύσκολο να γίνει αυτό, αν και ξέρουμε ότι έχουν αντικειμενικές ανάγκες και θέλουμε, θέλουν συγγνώμη, να τους βοηθήσουμε, να τις καλύψουν, αλλά και εμείς θέλουμε να έχουμε κάποιες διασφαλίσεις ότι όλα θα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες. Και κυρίως μας ενδιαφέρουν οι Σύροι στην Τουρκία, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός στόχος του μηχανισμού των προσφύγων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κιόλερ για 10 ε, λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη των Επιτροπών, θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος κύριος Ποπόφσκι. Όπως γνωρίζετε, στην Τουρκία υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Μιλάμε για καταγεγραμμένους πρόσφυγες. Δεν είναι όμως όλοι Σύροι. Ε, αυξάνεται ο αριθμός Ιρακινών, Ιρανών, Πακιστανών συγκεκριμένα Βέβαια, η ομάδα που μας απασχολεί περισσότερο είναι οι Σύριοι πρόσφυγες και εδώ μιλάμε για περίπου 3,6 εκατομμύρια καταγεγραμμένους Σύρους πρόσφυγες. Να τονίσω το καταγεγραμμένοι. Ο συνάδελφος μίλησε για τις δύο δόσεις της ε, διευκόλυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και ίσως σας ε, μπερδεύει κάπως αυτό, διότι εμείς σας λέμε ότι συνεχίζονται ε, τα προγράμματα, ότι υλοποιούνται αλλά ακούμε διάφορα παράπονα από την τουρκική πλευρά ότι δεν ε, έρχονται τα κονδύλια. Η δική μας απάντηση είναι καταρχάς ότι εμείς υλοποιούμε τα project ε, όσο μπορούμε, βοηθώντας ε, όχι την, το Ταμείο της Τουρκίας, αλλά τους πρόσφυγες μέσω διαφόρων διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, μέσω των ε, υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένων ΜΚΟ της ε, Τουρκίας καθώς και της ε, Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ρηθρού Σταυρού και των Συναφών Οργανώσεων. Αξιολογούμε και μετρούμε τις τα αποτελέσματα κοιτώντας τις δεσμεύσεις, κοιτώντας τις διάφορες συμβάσεις και τις εκταμιεύσεις. Οι εκταμιεύσεις αυτές φυσικά είναι εκταμιεύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια σε εταίρους με τους οποίους έχουν συναυθεί σχετικές συμφωνίες. Και νομίζω ότι μπορούμε να σας παρουσιάσουμε πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ε, το ελεκτικό συνέδριο άλλωστε διεξήγει τους ελέγχους και ε, αναφέρει ότι όλα βαίνουν καλώς. Οι εκταμιεύσει κονδυλίων και η υλοποίηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο της διευκόλυνσης αυτής είναι πέντε φορές γρηγορότερες από ότι ε, οι εκταμιεύσει για τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. σε ό,τι αφορά τώρα την ε, συμμόρφωση, θα μπορούσα να πω ότι σε γενικές γραμμές η υλοποίηση είναι, ε, γίνεται με με το σωστό τρόπο έχουν εκταμιευθεί το 100% των πρώτων τριών δισεκατομμυρίων της διευκόλυνσης και τώρα βρισκόμαστε στο 80% της ε, δεύτερης δόσης. Αναμένουμε το 100% στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Και αναμένουμε να ολοκληρωθεί η εκταμίευση μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, να αναφερθώ στο ότι μιλάμε μεν για την διευκόλυνση ως ένα σύνολο, όμως ε, αν κοιτάξουμε με μεγαλύτερη προσοχή θα δούμε ότι το 81% ε, των κονδυλίων διοχετεύεται σε ανθρωπιστική βοήθεια και το υπόλοιπο με αναπτυξιακή βοήθεια. Και ποια είναι η διαφορά εδώ. Η ανθρωπιστική βοήθεια από τη μία είναι πιο γρήγορη. Υπάρχει ε, πολύ γρήγορη διαδικασία εκταμίευσης, ανταπόκριση σε άμεσες ε, ανάγκες του ε, πληθυσμού. Βέβαια, να πω εδώ ότι δεν βρίσκονται όλοι οι πρόσφυγες σε κατάσταση ανάγκης. Η βοήθεια λοιπόν παρέχεται με βάση τις ε, άμεσες ανάγκες, δηλαδή σύντηση, στέγαση, συνθήκες υγιεινής. Έπειτα υπάρχει ο τομέας της εκπαίδευσης, της ε, κατάρτισης, σχολικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι τομείς οι οποίοι δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά της αναπτυξιακής βοήθειας. Σε ό,τι αφορά τώρα την, ε, την ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν δύο κύρια προγράμματα, εμβληματικά προγράμματα. Οι πληροφορίες φυσικά είναι διαθέσιμες στο κοινό, μπορείτε να τις ε, δείτε ή να συνομιλήσετε με μένα και με τους συναδέλφους για τις λεπτομέρειες, αλλά τα δύο εμβληματικά προγράμματα λοιπόν είναι από τη μία το δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας και η μεταφορά κονδυλίων για διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το δίχτυ τώρα κοινωνικής προστασίας παρέχει μηνιαίες πληρωμές άμεσα στους πρόσφυγες μέσω ε, καρτών. Εδώ εποφελούνται 1,7 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκία. Και τονίζω την Τουρκία διότι φυσικά σύμφωνα με τον κανονισμό για την σχετική διευκόλυνση παρέχεται το δικαίωμα και η υποχρέωση να χορηγείται βοήθεια στους πρόσφυγες στην Τουρκία. Γι' αυτό ο συνάδελφος όταν είπε ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ αναφέρθηκε σαφέστατα στο ότι δεν είμαστε σε θέση να στηρίξουμε την πλήρη ένταξη των Σύρων προσφύγων στη Συρία ως αποτέλεσμα των τουρκικών επιχειρήσεων στη χώρα. Αυτό δεν είναι μια πολιτική μονοδήλωση, αλλά και νομική, διότι η διευκόλυνση ε, νομικά δεν μας επιτρέπει να την χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 6 δισεκατομμύρια εκτός ε, τουρκικού εδάφους. Υπήρξε λοιπόν ε, μια πολιτική απόφαση να στηριχθούν οι Σύριοι πρόσφυγες στην ε, Τουρκία, αλλά και ε, ο νομικός χαρακτήρας της ε, διευκόλυνση δεν επιτρέπει τίποτα άλλο. Τώρα, να κάνω και μια πολύ σημαντική ανακοίνωση στο πλαίσιο αυτό. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώσαμε ότι από τον Απρίλιο του 2020 και μετά θα έχουμε και έναν νέο εταίρο που θα βοηθά στην υλοποίηση ένα, ε, το Παγκόσμιο Επιστημιστικό Πρόγραμμα είχε δραστηριοποιηθεί μέχρι τώρα, αλλά στο μέλλον θα αναλάβει τα ενία ο ερυθρό. Ε, Σταυρός. Η Τουρκία φυσικά είναι σημαντικός εταίρος, αλλά ο Ερυθρός ε, Σταυρός με τις όμως Ενώσεις τους είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην υλοποίηση του προγράμματος. Μέσω λοιπόν του Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε επικοινωνήσει και με το ηλεκτρικό συνέδριο και έχουμε λάβει την έγκριση για να χορηγούνται έτσι περισσότερα κονδύλια στους πρόσφυγες άμεσα χωρίς να χάνονται κονδύλια στη δίκηση. Μειώνοντας λοιπόν το κόστος και ε, αυξάνοντας τα ωφέλη για τους πρόσφυγες. Επίσης, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, χορηγείται βοήθεια σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Το πρόγραμμα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίω ε, ως προς τον προϋπολογισμό τους και περίπου μισό εκατομμύριο ε, παιδιά από τη Συρία μπορούν να έχουν λοιπόν εκπαίδευση η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, οι προκλήσεις. Από τη μία αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανάγκες. Όμως, συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη ΔΕΛΤΑ ΕΝΙΑΡ, για να δούμε πώς η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην κοινωνική ασφάλεια, αλλά και στον χώρο της εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, διεξάγονται οι συνομιλίες και δεν μπορούμε να σας πούμε ακόμα τι μελγενέστε λόγω των ε, συζητήσεων για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, βέβαια, καθώς παρατείνεται η κρίση, θα πρέπει να ε, εντείνουμε και εμείς ε, τις προσπάθειες ε, επίλυσης. Έπειτα, χρειάζεται και το κατάλληλο περιβάλλον για να μπορούμε να υλοποιήσουμε τα διάφορα project. Και αυτό σημαίνει πολλά πρακτικά ε, ζητήματα πρέπει να επιληθούν, δηλαδή να λαμβάνουμε τις σχετικές άδειες εξάσκησης επαγγέλματο, να ε, βελτιωθούν ορισμένες ε, λεπτομέρειες, να γίνει εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας. Πολλές φορές έχουμε προβλήματα στη συλλογή δεδομένων ακριβώς λόγω ε, το, της νομοθεσίας ε, προστασίας δεδομένων τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα επιληθούν τα ζητήματα αυτά σύντομα. Να σας πω επίσης ότι ε, με τις τουρκικές αρχές έχουμε μια αρκετά καλή συνεργασία για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Έτσι λοιπόν Αυτά ω προ τις εκταμιεύσει, Όπως σας είπα, έχει εκταμιευτεί το 100% της ε, πρώτης, ε, του πρώτου μέρου και το 81% του δεύτερου. Τώρα, έχω 13 δευτερόλεπτα, μπορώ να σας πω για τη Βόρεια ε, Συρία υπάρχει ένα πρόγραμμα 170 εκατομμυρίων ευρώ που είναι εκτός τη διευκόλυνση και αφορά μόνο τη Συρία. Στα βόρεια-ανατολικά της Συρίας όπου έχουν γίνει επιχειρήσει από την Τουρκία έχουν δοθεί γραμμα, ε, 68 εκατομμύρια ευρώ για ε, βοήθεια από αυτή και από άλλες γραμμές του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση κρίσεων. Υπάρχει όντως πρόβλημα. Πολλοί εργαζόμενοι στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εγκαταλείψει την περιοχή και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ε, βοηθήσουμε τους εκτοπισμένους. Οι επιχειρήσεις της Τουρκίας έχουν ε, προκαλέσει άλλους 100.000 εσωτερικά εκτοπισμένους σύρου. και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ε, ανταποκριθούμε στι ανάγκε που έχουν για στέγαση, σύντηση και υγιεινή. Και τώρα θα έχουμε το γύρο συζητήσεων που θα υποβάλλουν ερωτήσει, οι συντονιστές καταρχάς και μέλη μετά. Ο εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία θα πρέπει να μιλήσει, ο κ. Σάνσε Σταμόρ. Πρώτα απ' όλα όμως ξεκινήσουμε με ένα γύρο των συντονιστών. Έχουμε εδώ τρεις επιτροπές παρούσες, οπότε να έχουμε ένα συντονιστή για κάθε πολιτική ομάδα. Όχι όλους συντονιστές των τριών εμπλεκομένων επιτροπών. Ένας από κάθε μία. Ο κ. Γκέλλερ να ξεκινήσει. Θέλετε να μιλήσετε εκ μέρου του ΕΛΚ. Ε, δύο λεπτά το πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί σαφέστατα για τις ε, επιχειρήσεις της Τουρκίας σε Συριακό έδαφος. Υπάρχει μια συνένεση ευρεία για την στήριξη των ε, Σύρων προσφύγων ε, τόσο στη Συρία όσο και στην Τουρκία. Και είναι λογικό το, η διευκόλυνση αυτή να αφορά το τουρκικό έδαφος και όχι την Συρία, γιατί μιλάμε για πρόσφυγες. Τώρα, κύριε Γκάλερ, κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει η διερμηνία, υπάρχει, έχουμε. Πολύ ωραία, συνεχίστε. Ωραία, να, να πω πρώτα κάτι για να μεταφραστεί βέβαια και αυτό. Συνεχίζω λοιπόν ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενό διλήμματος. Ε, τι θα κάνουμε δηλαδή εάν ο Ερντογάν ε, δεν ε, συμπεριφερθεί σύμφωνα με αυτά που έχει υποσχεθεί. Εάν πάρει τους πρόσφυγες από, από τους καταβλισμούς προσφύγων και τους στείλει στα σύνορα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποια θα είναι η αντίδρασή μας σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει τις ε, συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι υπάρχουν πάρα, πολλά, πάρα πολύ ψηλά κονδύλια για την προενταξιακή βοήθεια. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, ο κύριος Ερντογάν έχει απειλήσει ότι θα ανοίξει τις πόρτες. Ξανά τις πόρτες προς ε, την Ευρώπη, έτσι ώστε να εκδικηθεί σε περίπτωση που υπάρξουν ε, κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτήν την πολύ συγκεκριμένη ε, επιλογή που ανέφερε ο κύριος Ερντογάν. Δεν βλέπω να είναι εδώ κυρία Τσίπελ που ζητούσε το λόγο. Πάμε στον επόμενο, για το Ρινιού, η κυρία Έντφελτ. Και αν εμφανιστεί η κυρία Σίπελ θα πάρει το λόγο. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ποπόφσκι και τον κύριο Κολάη. Δύσκολη κάπως αυτή η κουβέντα. Μιλάμε για χρηματοδότηση, για υποστήριξη των προσφύγων, στήριξη ανθρώπων και ταυτόχρονα πρέπει να συζητούμε και μεγάλα πολιτικά ζητήματα που έθιξε ο συνάδελφός μου από το ΕΛΚ. Τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να αναστείλουμε την υποστήριξη στον κόσμο και ταυτόχρονα η κατάσταση ίσως να αλλάξει. Όλα εξαρτώνται από τον κύριο Ντόγαν. Με τα χαρά σου άκουσα ότι είπατε ότι επουδενή δεν θα δώσετε οικονομική υποστήριξη σε διποτε επιστροφές που δεν είναι εθελοντικές. Πώς θα εξακριβωθεί αυτό όμως, ότι θα είναι εθελοντικές. Γιατί έχουμε αναφορές για κόσμο που επιστρέφει οι αρχές λένε ότι επιστρέφουν με τη θέλησή τους, ενώ αυτοί που επιστρέφουν λένε ότι δεν είναι καθόλου με τη θέλησή τους. Πώς θα το εξακριβώσουμε αυτό. Το θεωρώ άκρο ανησυχητικό. Και αισθάνομαι κάπως παράξενα, διότι θα πρέπει το πολιτικό θέμα να το θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα με το πρόγραμμα για την Τουρκία. Πάντα ήταν διστακτικό από την αρχή το Κοινοβούλιο. Δεν είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Αλλά ποια είναι η πολιτική βάση της διευθετήσεως. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση, όχι μόνο τις ότι θα κάνουμε αν συμπεράνουμε ότι δεν λειτουργεί πλέον το σύστημα και ότι εξαρτώμεθα απόλυτα από τη βούληση ε, του κυρίου Ερντογάν. Κυρία Σίπελ, δεν ήρθε ακόμα. Πράσινη, κυρία Τρίκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Στρίκ και τους, ε, ε, τους επιτρόπους για την παρουσίαση. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπε η κυρία Ιντφελτ. Ανησυχούμε πολύ για τη μοίρα των προσφύγων που διαμένουν στην Τουρκία τώρα. Με τα χαράς ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι αυτή η ζώνη ε, που δημιουργήθηκε στη Συρία είναι ασφαλής στην έκθεση προόδου όμως για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη μετανάστευση θέλουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξηθούν οι επιστροφές στην Τουρκία αντί να αυξηθεί η κατάσταση από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξακολουθεί να ισχύει αυτή η απειλή για απέλαση ανθρώπων που επιστρέφονται στην βορειοανατολική Συρία. Άρα, ερώτημα, σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διατείνεται ακόμα ότι είναι ασφαλής τρίτη χώρα η Τουρκία και να πιστεί έτσι η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τις διαδικασίες ασύλου για, τη, για τους Σύρους πρόσφυγες. Και αυτές οι αναφορές που έχουμε για τις κατα... αναγκαστικές επιστροφές στη Βόρεια Συρία, πώς μπορούμε να εξακριβώσουμε τι συμβαίνει, ότι είναι μόνο εθελούσιες επιστροφές και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν γίνονται αναγκαστικές επιστροφές. Και αν ξεκινήσει την απέλαση ε, αυτών των ανθρώπων η Τουρκία, εμεί τι θα κάνουμε. Και τώρα πάμε στο ID. Ο κύριος Μαριάννη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα τις παρουσιάσεις των δύο εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κύριου Κέλλερ και του κυρίου Ποπόφσκη. Κύριε Ποπόφσκη, μιλάτε για την σωστή ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην Ευρώπη. Ο άλλο εκπρόσωπο αναφέρθηκε στο πρόγραμμα για την Τουρκία. Θέλω να πω ότι συμμερίζομαι τι ίδιε ανησυχίε όπω και εκπρόσωποι των τριών άλλων ομάδων που τοποθετήθηκαν. Στην πραγματικότητα, τι συμβαίνει. Δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα όσον αφορά το πρόγραμμα και τα ποσά που δίδονται στην Τουρκία. Η ομάδα μα το κατήγγειλε επανειλημμένα αυτό. Είμαστε όμοιροι πολιτικοί των εκβιασμών του κ. Ερντογάν. Τίθεται σήμερα το εξή ερώτημα αν πρέπει να επεξετάσουμε την πολιτική μας σε αυτή την περιοχή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα είναι η στάση μας δηλαδή έναντι της κυβερνήσης της Τουρκίας και ο καλύτερος τόπος να εγκατασταθούν οι Σύριοι πρόσφυγες δεν είναι στην Ευρώπη, δεν είναι στην Τουρκία, είναι στη Συρία. Αν είναι θελοντικέ όμω οι επιστροφέ. Αν είναι θελοντικέ. Σήμερα η κατάσταση στη ποια είναι, ότι στη Συρία με την εξαίρεση του θύλακα του Ιντλίμπ ε, επικρατεί ειρήνη στην περιοχή. Μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο, πιο ανθρώπινο και λιγότερο δαπανηρό σήμερα να δούμε αν μαζί με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις μπορούμε να συνεργαστούμε για την επιστροφή των σύρων προσφύγων στα σπίτια τους. Διότι αν τελικά οι πρόσφυγες επιστρέψουν στις πατρίδες τους είναι πολύ καλύτερη λύση. Ευχαριστώ κύριε Μαριάννη για το ECR. Η κυρία Σκύμπα. Όχι. Ναι, ναι. Η κυρία Κέμπα. Είμαι εδώ, λέει η κυρία Κέμπα. Εδώ, εδώ είμαι. Ορίστε, ορίστε, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Κέμπα. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση είναι σοβαρότατη κατά την άποψή μου. Πρέπει να την εξετάσουμε από δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα έχουμε διπλωματικά θέματα και είναι πολύ σοβαρό το έργο της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Αντιμετωπίζουμε, βλέπετε, απειλέ από τον κύριο Ερντογάν. Μας εκβιάζει ο Ερντογάν. Απ' την άλλη, αντιμετωπίζουμε μια τεράστια απειλή που στρέφεται κατά των πολιτών, κατά των προσφύγων, κατά εκείνων που προέρχονται από τη Συρία ή των εσωτερικά εκτοπιστέντων διότι οι επιθέσεις στη Βόρεια Συρία δημιούργησαν και άλλες ε, μετακινήσεις ανθρώπων. Έχουμε ΜΚΟ εκεί που μας λένε ότι είναι τραγική κατάσταση εκεί, στο Χόλμς και στο Χαλέπι και επιδεινούται η κατάσταση και έχουμε όλο και περισσότερους εσωτερικά ε, εκτοπισμένους. Όσον αφορά αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να την αυξήσουμε, πιστεύω διότι είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι σωστό. Όσον αφορά τα άλλα είδη βοηθείας, όπως είναι αναπτυξιακή βοήθεια, αυτό είναι σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της Τουρκίας και άλλων χωρών. Ίσως πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Γιατί είναι τόσο σοβαρή κατάσταση. Πρέπει να πω ότι η Τουρκία, όπως είπε και η Νάντια Μουρατ πρόσφατα, ότι η Τουρκία επιτίθεται κατά των χωριών των Γιαζίδη και των γυναικών των Γιαζίδη ε, ε, που είναι θύματα του Ισλαμικού κράτους. Λοιπόν, η κατάσταση επιδεινούται. Αν λάβουμε υπόψη λοιπόν τι γίνεται στην Ιορδανία και στο Λίβανο, ότι και αυτές οι χώρες σχεδιάζουν επίσης να στείλουν τους Σύρους πρόσφυγες πίσω στη Συρία Λοιπόν, θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή στη Μέση Ανατολή και θα πρέπει να τη δούμε και στα πλαίσια της διπλωματίας. Για την ΚΟΕ, ο κύριος Ρουμπάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω συντονιστής ε, από την ΔΕΒΕ και από τη ΛΥΜΠΕ. Δύο ερωτήσεις ε, θέλω να θέσω. Η Επιτροπή θεώρησε ότι ε, θα εξαρτήσει την χρηματοδότηση της Τουρκία από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή θα κοιτάμε από την άλλη πλευρή ενώ επιτίθεται στη Ροτζάβα η Τουρκία και προβαίνει σε εθνοκάθαρση προκειμένου η τουρκική κυβέρνηση να συνεχίζει να αστυνομεύει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη η ερώτηση. Θα κοιτάμε από την άλλη ή θα εξαρτήσουμε από τους εμπισμούς των δικαιωμάτων τη χωρίς της βοήθειας. Ε, δεύτερον, έχοντας ε, κατά νου ότι η θα εξαρτησουμε απο τους Ευρωπαϊκούς δικαιωματων τη χωρις της βοηθειας δευτερον εχοντας κατα νου οτι αρχη της ε, με επιστροφής και καταγγέλουν οι ΜΚΟ, ε, 340.000 ε, Σύριοι καταγγέλλεται ότι έχουν επιστροφή χωρίς τη θέλησή τους ενώ υπόθηκε ότι ήταν θελούσιες επιστροφέ. Όμω εδώ έχουμε την έκθεση τη Διεθνού Αμνηστία, ε, όπου αναφέρονται αυτά τα δεδομένα. Ε, μπροστά σε αυτές τις, επιτροπές, ε, σε αυτές τις επιστροφές η Κομισιόν θέλει να υπενθυμίσει στα κράτη-μέλη να μην θεωρούν την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα. Πρόκειται για μια έκθεση τη Sea-Watch που έχουμε εδώ και έλεγε ακριβώς ότι η Κομισιόν συνέστηνε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρούν την Τουρκία μια ασφαλή τρίτη χώρα. Η Τουρκία όμως δεν είναι. Εσείς ε, πρόκειται να συστήσετε ε, να μην είναι ασφαλή τρίτη χώρα η Τουρκία και ε, τώρα θα ασχοληθείτε με αυτά τα θέματα που σας αναφέρω για τα οποία υπάρχουν αποδείξεις. Βλέπουμε ότι η κυρία Σίπελ επέστρεψε. Αν θέλετε το λόγο για δύο λεπτά για την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι πολλοί άσκησαν κριτική από την αρχή στη συμφωνία αυτή με την Τουρκία. Μία θετική πτυχή που ίσως ε, να υπήρχε στη συμφωνία αυτή, κατά την άποψή μου, θα ήταν να είχαμε χρόνο να προετοιμάσουμε καλύτερα τα δικά μας συστήματα για το πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των προσφύγων, να ενδυναμώσουμε τα συστήματά μας όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια ταχεία ε, και σωστή διαδικασία χωρίκησης ασύλου, αλλά να είμαστε και σίγουροι ότι μπορούμε να υποδεχτούμε ορθά τους πρόσφυγες και να ε, διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να στείλουμε πίσω ανθρώπους στις χώρες προέλευσης σε περίπτωση που δεν διώκονται εκεί. Όμως, από ό,τι βλέπω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιεί το χρόνο αυτό για να ενισχύσει τα συστήματά της. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και δίνουμε την εντύπωση ότι δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τη ε, μετανάστευση, ούτε την νόμιμη μετανάστευση, ούτε το θέμα της χορηγή ασύλου και είμαστε στα χέρια ενό ανθρώπου όπω ο Ερντογάν για να διασφαλίσει ότι δεν έρχονται πολλοί στην Ευρώπη. Και ξεχνάμε εντελώς το ότι οι περισσότεροι πρόσφυγες δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε έρχονται στην Ευρώπη. Μένουν σε άλλες χώρες γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, από την άποψη αυτή, αναρωτιέμαι από όλα τα ωραία λόγια που ακούμε επανειλημμένα για αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία. Υπάρχει πράγματι καλός λόγος να συνεχιστεί και ποιες προσπάθειες θα καταβάλλετε εσείς από την πλευρά σας για να υποστηρίξετε την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το τι καινούριο θα μπορούσε να υπάρχει για αυτό το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Και δύο τελευταία λεπτά. Ο κύριος Σάντσε Αμόρ, ο εισηγητής για την Τουρκία. Η ευρωπαϊκή πολιτική με την Τουρκία θα πρέπει να απαντήσει στην πολυπλοκότητα της σχέσης και θα πρέπει να έχει κατά νου τις ε, τάσεις και τις συγκυρίες. Ε, η τάση είναι ότι έχουμε προοδευτική απομάκρυνση και λήψη εμπιστοσύνης ε, που βασίζεται στις αυταρχικές τάσεις του καθεστώτος. Δεν μπορούμε να σε χρησιμοποιήσουμε την δικαιολογία για την Τουρκία, την απόπειρα πραξικοποιήματος για τις πολιτικές που εφαρμόζονται και επίσης η συγκυρία έχει να κάνει με το τεράστιο λάθος που αποτελεί αυτή η μονομερής επέμβαση στη Συρία. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου πράγματα που συμβαίνουν στην εγχώρια εσωτερική πολιτική της Τουρκίας. Ε, έχουμε την διπλή νίκη στην Κωνσταντινούπολη της αντιπολίτευσης και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην ανάλυση μας. Τα Ηνωμένα Έθνη μόλι το έκαναν, αναγνώρισαν το ρόλο της Τουρκίας ε, να διατηρεί στο εδαφός της αυτή τη τεράστια, το τεράστιο αριθμό προσφύγων. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε πολιτικές εντός της Ευρώπης με όλους αυτούς τους πόρους. Μήπως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Το θέμα είναι ότι ο μηχανισμός, το Ταμείο, ουσιαστικά είναι η μόνη εξομαλυμένη σχέση που έχουμε με την Τουρκία και η μοναδική και ο μοναδικό ε, τρόπος να βοηθήσουμε αυτά τα εκατομμύρια προσφύγων. Όχι ε, μέσω ένεση στην, στην τουρκική οικονομία. Γιατί μερικές φορές περνάει το μήνυμα ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στην τουρκική οικονομία. Όμως ε, πολύ λίγα πηγαίνουν στη δημόσια δίκηση στην Τουρκία. Το είπαν σχεδόν όλοι πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ούτε ένα ευρώ να μην χρησιμοποιηθεί άμεσα ή έμεσα για να διευκολύνει την επαναγκατάσταση που θέλει ο κύριος ε, Ερντογάν ε, στη Βόρεια Συρία ε, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα σε αυτή την ήδη πολύπλοκη δημογραφία όπως είπε ο Αντώνιο Γκουτέρες και όπως είπε το Κοινοβούλιο η μόνη επαναγκατάσταση που γίνεται πρέπει να είναι εθελούσια και αξιοπρεπής. Τώρα, ο μόνο τρόπο να τη διαχειριστούμε τη συζήτηση είναι ο εξή. Υπάρχει ένα σύντομο κατάλογος και τον κλείνουμε. Ένα λεπτό ο καθένα και κατόπιν θα έχουμε τέσσερα λεπτά για τι απαντήσει για τον κάθε μιλητή στο πάνελ. Θα πρέπει να περιμένει ο Έλληνα Υπουργό, αλλά όχι και υπερβολικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ο κύριο Μαυρίδη, παρακαλώ. Minute, maximum. Ναι. Έχουμε αυτές τις συζητήσεις. Η απάντηση από τους ε, εισηγητές είναι πολύ απλή. Αν δεν ήταν οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Το ερώτημα είναι ότι κάθε φορά που έχουμε την ίδια συζήτηση, τα πράγματα είναι χειρότερα. Η απάντηση για μένα είναι πολύ απλή. Απλώς φοβάμαι ότι αρκετοί εδώ δεν είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε ως έχει την πραγματικότητα. Λοιπόν, είμαστε ενώπιον ενός Ερτογάν, ο οποίος είναι ένας εγκληματίας κατά της ανθρωπότητας. Τόλμησαν να το πούν πολλοί άλλοι, όπως η Κάρλα Τεπόντε και πολλοί άλλοι διεθνώς αναγνωρισμένοι ερευνητές. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Δίνουμε χρήματα στον Ερτογάν και ο ίδιος ταυτοχρόνως προκαλεί νέους πρόσφυγες στη Βόρεια Συρία. Δεν θέλω να είμαι μέρος ενός τέτοιου εγκλήματος. Mr. Papadakis. Κύριε Παπαδάκη. Minute, maximum. Ένα λεπτό. Here. Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Ε, Ευχαριστώ. Νομίζω πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι ο κύριος Ερτογάν εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι εμείς πώς αντιδρούμε σε αυτούς τους εκβιασμούς. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε λέγοντας ότι εμείς πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες. Thank you, Mr. Furlas. Εδώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να απαντήσω στο ερώτημα των συναδέλφων αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερτογάν. Η Τουρκία απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγε αν δεν τον ικανοποιήσουμε. Η Τουρκία εισέβαλε σε ξένη χώρα και απειλεί τώρα να αλλάξει τη δημογραφική δομή αυτό που ονομάζει ζώνη ασφαλεία. Η Τουρκία εισέβαλε πριν 45 χρόνια και κατέχει ευρωπαϊκό έδαφο, την Κύπρο. Η Τουρκία πριν από μερικού μήνε μπήκε σε θαλάσσια περιοχή που ανήκει σε ευρωπαϊκό κράτο, είναι εκεί και μιλούμε για ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή επικράτεια. Και διαρωτόμαστε σήμερα εδώ ακόμα αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερτογάν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very... Καταρχήν, ε, να πω σε είπαν και κάποιοι συνάδελφοι για το θέμα της επαναγκατάστασης. Πώς ε, γνωρίζουμε ότι δεν ε, γίνεται με το ζόρι. Επίσης, ξέρουμε ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο για να προβεί σε δημογραφική μηχανική σε αυτή την εμπόλεμη κατά την απόψή μου ζώνη. Και η δεύτερη ερώτηση, το δεύτερο θέμα, έχει να κάνει με τα οικονομικά, με τα κονδύλια που δίνονται για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Έχουμε μια έκθεση του λεκτικού Συνεδρίου του 2018, όπου δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν ε, για το πώ ε, ένα δισεκατομμύριο ευρώ ξοδεύτηκαν και αν ξοδεύτηκαν για του ήρου πρόσφυγε. Ήθελα να συγκρίνουν οι ελεκτέ ε, την τον κατάλογο των προσφύγων της Τουρκίας με τον ε, κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν ε, τα χρήματα, όμως ε, τους αρνήθηκε πρόσβαση το Υπουργείο Κοινωνικής Μέριμνας της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν η ερώτησή μου βασικά είναι πώς ξέρουμε ότι τα χρήματα πήγαν εκεί όπου μας είπαν. Ευχαριστώ κύριε Προκατσίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν, θέλω να υπογραμμίσω την υποκρισία που διέπει το όλο ζήτημα και προκύπτει από το λάθος του να εμπιστευτούμε τα έλεγχο των ευρωπαϊκών συνόρων σε τρίτα κράτη. Και άκουσα ότι δεν υπάρχει έγχυση κονδύλιων ε, στα ταμεία της ε, τουρκικής κυβέρνησης. Δεν είναι αλήθεια όμως. Έχουμε τουλάχιστον τρεις συμφωνίες ε, με κυβερνητικά όργανα της Τουρκίας που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν αυτήν θα πρέπει να μου εξηγήσει κάποιος ε, γιατί ε, γίνεται ε, τελικά δίνεται αυτή η βοήθεια στην Τουρκία και όχι παραδείγματο χάρη στην Τινησία σαν να ε, ήταν μια λιγότερο ασφαλής χώρα από την Τουρκία που φτάνει η πλειονότητα των μεταναστών σήμερα ε, μέσω της Μεσογείου. Η αλήθεια είναι ότι μας εκβιώσουν γιατί τελικά πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιον άλλο να κάνει τη δική της δουλειά. Ευχαριστώ κύριος Γουάλλας. Ευχαριστώ. Είπατε ότι ο μηχανισμός ε, δεν θα επέτρεπε τα χρήματα νόμιμα να χρησιμοποιηθούν ε, για την κατάσταση σύρων προσφύγων στη Συρία. Δεδομένου ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η ιδέα ε, της Τουρκίας να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στη Βόρεια Συρία και όχι στην Τουρκία φαίνεται ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ανοιχτή φυλακή σαν τη Γάζα. Δηλαδή, αν θα βάλουμε πρόσφυγες ε, και θα βάλουμε πρόσφυγες ε, αργότερα σε αυτή την περιοχή. Μήπως ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε την κατάσταση στην ίδια Τουρκία για να διευκολύνουμε την επιστροφή πολλών προσφύγων. Μήπως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να έρθουν οι κυρώσεις κατά της Συρίας. Δεν έχει νόημα να έχουμε τις κυρώσεις κατά της Συρίας. Ε, οι περισσότεροι τζιχαντιστές έχουν εκδιωχθεί. Οι περισσότεροι Σύριοι θα επέστρεφαν αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε τη Συρία να σταθεί ξανά στα πόδια της. Μάλιστα, κύριε Σόφτκο. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση των προσφύγων. Και αυτό είναι το θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τα μέσα να πολεμήσει τον Ερντογάν αλλά θα πρέπει να σταματήσουμε τη ροή των προσφύγων στα Βαλκάνια. Uh, Γιατί θα ανοίξουν άλλες πληγές. Θα δημιουργηθούν κάποιοι μηχανισμοί μαζί με τους τόπιου πληθυσμούς ε, για την ένταξη των προσφύγων. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, τόσα εκατομμύρια έχουμε εκατομμύρια πρόσφυγες ε, και οι τοπικές κοινότητες τους απορρίπτουν. Ποιο είναι το νόημα λοιπόν να έχουμε όλους αυτούς τους πρόσφυγες ε, και πόσα χρήματα θα δαπανηθούν ε, σε ντόπιε υποδομές. Γιατί μας λένε ότι αυτό δεν γίνεται. Αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν λοιπόν στο χαμηλότερο επίπεδο προκειμένου να ενταχθούν οι πρόσφυγες και όχι να μένουν σε καταβλησμούς τόσα χρόνια δεν νομίζω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Ερντογάν. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις τοπικές κοινότητες προκειμένου να βοηθήσουν του πρόσφυγε αυτού να ενταχθούν. Ευχαριστώ κύριε Ζημιούκ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Στην Ευρώπη κλείνουμε τα μάτια μας στις διαπραγματεύσεις με τον Ερντογάν. Τον θεωρούμε εταίρο, όμως δεν είναι εταίρος, είναι αντίπαλός μας. Χρησιμοποιεί εμάς για τα δικά του συμφέροντα και ε, μαχαιρώνει πλησόπλατα τόσο εμάς όσο και τους ε, πρόσφυγες. Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί ένα τέλος εκεί, να ρίξουμε την προσοχή μας στη Συρία και να διαπραγματευτούμε με τον Ασάντ. Χρειάζεται λοιπόν να έρθουν αυτές οι κυρώσεις για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους επί τόπου. Αυτό είναι προς το συμφέρον πιστεύω όλων. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπέ έχει λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι αντιμετωπίζουμε επανειλημμένα ε, τις πιέσεις ε, διάφορες επιθέσεις στην κατάκτηση της Κύπρου, την επίθεση που έκανε κατά της Συρίας, ε, επίθεση στη Συρία κατά των Κούρδων. Και συνέχεια τους πληρώνουμε 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τα θέματα που μεταστατικά δίνουμε στην, Τουρκία και δεν συμμορφούνται η Τουρκία από την αρχή έχουμε δώσει περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σταματήσουν οι εκβιασμοί του Ερντογάν να πληρώνουμε την Τουρκία. Πρέπει να σεβαστούμε την εδαφική κυριαρχία της Συρίας και όπως είπαν οι συνάδελφοι όπως Μαριάννη να εστιαστούμε στα 3,6 εκατομμύρια Σύρους που είναι ε, στην Τουρκία να επιστρέψει στη Συρία χωρίς να αποφασίσει τον Ερντογάν που θα πάνε σε μια ζώνη που θέλει να ελέγχει μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Ευχαριστώ. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Παρακαλώ προσπαθήστε να, είστε, να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Και έχουμε και Επιτροπή ΑΦΕΤ που θα συνεδριάσει τώρα στις 10. Και έχουμε τον Έλληνα Υπουργό που μας περιμένει. Αν έχει μείνει κάτι να πείτε, στείλτε το γραπτός και μπορούμε να διανύουμε τις ε, απαντήσεις. Παρακαλώ ένα τετράλεπτο ο καθένας αν έχετε την καλοσύνη. Ο κ. Ποπόφσκι πρώτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Πρώτα είναι ο άνθρωπος. Εστιαζόμεθα επί των σύρων που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και θέλουμε να συνεχίσουμε τη βοήθειά μας για αυτούς. Δεν θα υποστηρίξουμε σίγουρα τη μετεγκατάσταση, την αναγκαστική απομάκρυνσή τους που του στέλνουν στη Συρία, είτε από την Τουρκία, είτε από το Λίβανο, είτε από άλλη χώρα. Αν αποφασίσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν, θέλουμε να μα διαβεβαιώσει η πατιαρμοστία του ΟΗΕ ότι όλα γίνονται σύμφωνα με του κανόνε. Αυτέ οι επιστροφέ θα πρέπει να είναι αξιοπρεπεί Εθελούσια. Ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτιέρε, συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ετογάν πριν από τρει ημέρε, συζήτησαν το θέμα δεν ξέρουμε ακόμα κατά πόσον η τη του ΟΗΕ θα έχει πρόσβαση στη Βόρεια Συρία. Την περασμένη φορά που το εξέτασα, την περασμένη Παρασκευή, δεν είχε κάτι τέτοιο. Αλλά πραγματικά πρέπει να μας διαβεβαιώσει η πατιαρμοστία ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα των ε, επιστρεφόντων. Έχουμε κάποια μέτρα παρακολούθησης καταστάσεως, πώς δαπανούνται τα χρήματα σε ποιον πηγαίνουν τα χρήματα. Το συζητούμε τακτικά με τα κράτη-μέλη μας αυτό και με την Τουρκία. Και επόμενη ευκαιρία θα είναι η Ευθύνους Επιτροπή για το Μέσο Διευκόλυνσης στις 9 Δεκεμβρίου. Και ελπίζουμε ότι ο πρόεδρος της ΑΦΕΤ και τα μέλη του Κοινοβουλίου θα είναι παρόντα. Θα στείλουμε πρόσκληση σύντομα για αυτή την εκδήλωση. Καλή ευκαιρία να συζητηθεί η κατάσταση, η επιτόπια Γνωρίζω ότι αυτό το θέμα της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας είναι κάτι που έχει τεθεί επανειλημμένος. Οι διεθνείς αρχές κρίνουν, σε αυτές βασιζόμαστε επί της Ελλάδος πιο συγκεκριμένα. Δίνουμε υποστήριξη ταυτόχρονα σε εκείνους που έχουν μετεκατασταθεί στην ε, Τουρκία, νόμιμη βοήθεια, χρηματοδοτούμε, νομική βοήθεια μάλλον χρηματοδοτούμε και δεν θέλουμε να επιδεινωθεί κατά στην Τουρκία που αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Όσον αφορά τη συνεχιζόμενη συζήτηση για το σύστημα ασύλου στην Ευρώπη, πράγματι η πρόεδρο, η νέα πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ανακοίνωσε, θέλει να ετοιμάσει ένα σύμφωνο για το ασύλο στην ε, Ευρώπη. Θέλω να προδικάσω τι θα κάνει η νέα πρόεδρο όταν θα ξεκινήσει η νέα θητεία τη. Αλλά είναι από τι πρώτε προτεραιότητε τη. Το ανέφερε τον Ιούλιο, όταν μίλησε εδώ στο Κοινοβούλιο. Στο Στρασβούργο, μάλλον. Στο Κοινοβούλιο. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πού πηγαίνουν τα χρήματα. Το ανέφερε ο εισηγητής. Πράγματι δαπανούμε τα περισσότερα από τα 6 εκατομμύρια μέσω των εταίρων αναπτυξιακών φορέων, ΜΚΟ, τραπεζών, ερυθρού σταυρού. Έτσι θέλουμε να παραμείνει η κατάσταση. Τα χρήματα που πηγαίνουν στα τουρκικά υπουργεία δεν είναι δημοσιονομική υποστήριξη. Του επιστρέφουμε στα πάνε, ό,τι ξοδεύουν για σχολεία, κλινικέ, του αποζημιώνουμε. Αλλά δεν είναι ρευστό που, που καταβάλλεται γρήγορα. Δεν θα υποστηρίξουμε κάποια κοινωνική αλλαγή αναγκαστική στη Συρία, αλλαγή των πληθυσμών. Σαφής προσέγγιση αυτή και η θέση των ΗΠΑ ακριβώ η ίδια. Είμαστε ενωμένοι Όσον αφορά την ένταξη των προσφύγων, κάνουμε πολλή δουλειά στην Τουρκία. Επενδύουμε σε υποδομές, επαγγελματική κατάρτιση και παιδί κατάσταση στη Βοσνία είναι κάπως διαφορετική. Εκεί η βασική μας προσπάθεια να βελτιώσουμε τις δυνατότητες υποδοχής. Και δαπανίσαμε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για ειδικά μέτρα στη Βοσνία. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και θέλουμε να παρέμβουμε. συνήθω είναι αργή ρυθμή που κινούνται τα πράγματα στη Βοσνία και δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σκέλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα πλούσια αυτά σχόλια. Επιγραμματικά, η ασφαλή επιστροφή των προσφύγων. Έχουμε κάποια κριτήρια που εφαρμόζουμε σε όλο τον κόσμο και σε αυτή την κρίση. Η επιστροφή των προσφύγων στην πατρίδα του πρέπει να είναι αξιοπρεπή, εθελούσια, ασφαλής, βιώσιμη. Όχι να μπαίνουν και να ξαναβγαίνουν. Ποιο θα το παρακολουθεί αυτό, ένα οργανισμό πλήρωνται γι' αυτό, είπα τη αρμοστία του ΙΕ τη προσφυγέ. Πρώτη στο θέμα, αν θέλουμε αξιοπρεπή, εθελούση, ασφαλή και βιώσιμη επιστροφή στη Συρία, είναι, είπατε, αρμοστία να λειτουργεί ελεύθερα στη Συρία. Αυτό δεν γίνεται σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό θα είναι λογικό, αν οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν αυτό που ανακοίνωσαν θέλουν να κάνουν, είναι να φροντίσουν, ούτω ώστε είπατε αρμοστία του ΙΕ να μπορεί να κινηθεί εκεί, να λειτουργήσει εκεί. Η κυρία Σίπελ υπενθύμησε ότι οι περισσότεροι πρόσφυγε σε όλο τον κόσμο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Σύμφωνα με εκτιμήσει, έχουμε 70 εκατομμύρια ανθρώπου οι οποίοι έχουν ε, μετακινηθεί υποχρεωτικά, αναγκαστικά σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι είναι μετανάστε, αλλά 25 εκατομμύρια από αυτού είναι πραγματικοί πρόσφυγε. Έχουμε 1,8 δι ευρώ για να καλύψουμε του πραγματικού πρόσφυγε. Τα περισσότερα χρήματα χρησιμοποιούνται για ανθρωπογενεί κρίσει. Ανθρωπογενεί κρίσει οδηγούν σε αναγκαστική ε, μετακίνηση των πληθυσμών. Χρειάζεται να κάνουμε περισσότερο να υποστηρίξουμε, όπω αναφέρθηκε. Ναι, αγαπητά μέλη τη Επιτροπή, ε, μάλλον τον φορέα του προπολογισμού, δώστε μα περισσότερα χρήματα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Άλλη ερώτηση για την προστασία των δεδομένων και πρόσβαση στα δεδομένα. Πράγματι, είπα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση που αφορά την πρόσβαση δεδομένα, όσον αφορά του πρόσφυγε εντό τη Τουρκία σημειώνεται πρόοδο και ερχόμαστε σε νέα συμφωνία με του Τούρκου πάνω σε αυτό. Αυτό τακτικά το θέτουμε σε συνομιλίε ψηλού με του Τούρκου. Αυτή τη στιγμή όμω δεν θα ήταν δίκαιο να πούμε ότι δεν έχουμε ιδέα για το τι συμβαίνει. Εργαζόμαστε βάσει δειγματοληψία, βάσει πληροφοριών από του διαφόρου φορεί με του οποίου συνεργαζόμαστε. Έχουμε, θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία και αυτό το διαπραγματευόμαστε. Κάποιο βουλευτή είπε γιατί δεν έρονται οι κυρώσει κατά των Συριακών αρχών. Και όλα θα πήγαν καλά αντί αυτή την περίπτωση. Εγώ έχω αμφιβολίε να μην λησμονούμε ότι 80% τουλάχιστον εκείνων που έφυγαν από τη χώρα του, από την Συρία, δεν προσπαθούν να ξεφύγουν από το Ισλαμικό κράτο, από τον Ντάε. Προσπάθησαν να βρουν καταφυγή από τι γειτονικέ χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των φρικαλαιοτήτων του καθεστώτο Ασάντ. Και αν θέλετε την κατάσταση Ιορδανίας, να την πάτε σαν παράδειγμα, στην Ιορδανία τα τελευταία τρία χρόνια 35.000 Σύριοι πρόσφυγες επέστρεψαν στην Συρία. Αλλά 650.000 παραμένουν στην Ιορδανία. Και ακόμα και αν η Τουρκία εφάρμοζε επιστροφές του Σιπίν στη Συρία, μεγάλος αριθμός Σύρων προσφύγων είμαι σίγουρος ότι θα παρέμενε στην Τουρκία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επενδύσουμε πολύ σοβαρά, δεν θα έλεγα στον αφορά αλλά τουλάχιστον να δούμε πώς μπορούν να ζουν. Παιδεία, συμμετοχή στον οικονομικό βίο της ε, χώρας οικοδεσπότου. Να βοηθήσουμε την οικονομία της χώρας που είναι οικοδεσπότης και αυτοί να ζουν πιο αξιοπρεπή ζωή. Είναι δέκα φορές πιο αξιοπρεπές να κερδίζεις τα δικά σου λεφτά από το να εξαρτάσαι από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τρόφιμα σου δίνει. Όλο και περισσότερο στην Τουρκία, στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στο Ιράκ η Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡ και ΕΚΟ επενδύουν στην υποστήριξη του βίου των ανθρώπων αυτών, να μπορούν να βγάλουν χρήματα, να εργαστούν μέσω επαγγελματική κατάρτιση, να βοηθήσουμε να δημιουργήσουν δικέ επιχειρήσει. Αυτό συμβαίνει, αλλά βέβαια γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο και να έχουμε φορεί οι οποίοι αποδέχονται ότι αυτοί οι πρόσφυγε δεν πρέπει να παραμένουν σε στρατόπεδα και καταβλισμού, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν πλήρω στην οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Ας ακούσουμε όμως ε, τα τελικά σχόλια των ε, Προέδρων των άλλων Επιτροπών. Αρχίζω με τον ε, κύριο Τομπίας Τζοεφ. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται από αυτά που ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο και περίπλοκο ζήτημα, το οποίο είναι και πολιτικό. Χρειάζεται λοιπόν να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η Τουρκία είναι η χώρα που υποδέχεται τους περισσότερους πρόσφυγες στον κόσμο. Αυτό για μας είναι πολύ βασικό στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Όμως από αυτή την σύντομη ανταλλαγή απόψεων συμπεραίνω ότι χρειάζεται καλύτερος έλεγχος της κατάστασης, όχι μόνο έλεγχος ε, των κονδυλίων και πώς αυτά χρησιμοποιούνται, αλλά έλεγχος της υλοποίησης ε, και της εφαρμογής των προγραμμάτων και των δικών μας πολιτικών. Χρειάζεται λοιπόν μια σαφής δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Εδώ ολοκληρώνεται το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Τώρα η κάθε επιτροπή θα συνεχίσει με τη δική της ημερήσια διάταξη. Εμείς ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα παραμείνουμε εδώ έτσι ώστε να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης όπου θα υποδεχτούμε τον Έλληνα Υπουργό.